Ε, Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ε, είμαι η Αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και έχω την τιμή να συμπροεδρεύω ε, σε αυτήν την κοινή επιτροπή γυναικών, γυναικών και επιτροπής νομικών υποθέσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που έχουμε μαζί μας, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την ε, φίλη και συνένοχο υπουργό του Λουξεμβούργου Λίδια Μίσ, ε, για να συζητήσουμε ε, για το θέμα της ε, αντιπροσώπευσης των γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων. Δεν έχω κανένα ε, λόγο να σας ε, θυμίσω πώς έχουν τα πράγματα και ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζω ότι αποτελεί προτεραιότητα το θέμα αυτό ε, για την Λουξεμβουριανή Προεδρία και μάλιστα η Υπουργό είναι δεσμευμένη απέναντι στο θέμα αυτό να το συζητήσει και να το αντιμετωπίσει. Είμαι ευτυχής επίσης ε, να, που θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε την κυρία Ντυρό και να μας ε, ε, μιλήσει για τις συστάσεις ε, του ε, Θα δώσω όμως το λόγο στην συμπρόεδρό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κυρία Συμπρόεδρε και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που συμπροεδρεύω σήμερα το απόγευμα σε αυτήν την κοινή συνεδρία στον Επιτροπ... της Επιτροπής μας με την Επιτροπή των... την Γιούρη. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει το Νοέμβριο του 2013 το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε ε, και είναι μάλιστα σωστό και ισορροπημένο ε, όσον αφορά δηλαδή αυτήν την ισόρροπη αντιπροσώπευση των γυναικών ε, στις, στα Συμβούλια των Επιχειρήσεων. Πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε, παλεύουμε για το θέμα αυτό, αλλά εδώ πραγματικά θα προσθεθεί ένα πολύ σημαντικό input και θα δώσουμε νέα ορμή στο θέμα. Ε, και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και η Προεδρία του Λουξεμβούργου ε, στήριξαν αυτήν την συμφωνία και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί έχουμε κάνει πολύ καλή ομαδική δουλειά. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι εύκολα και η στιγμή δεν είναι εύκολη. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αγωνιστεί για να επιτύχει συμφωνία ξεκινώντας από την επόμενη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις του Συμβουλίου αυτά που έχει να μας πει σήμερα. Γνωρίζουμε ε, ότι το Συμβούλιο δεν ε, είναι έτσι πολύ ε, θερμό όσον αφορά αυτήν την σύσταση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες είναι λίγο χλιαρές όσον αφορά ε, αυτό το ζήτημα. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μας να ε, επιστρέψουμε στις χώρες μας και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας έτσι ώστε να ξέρουμε ποιο θα είναι το μήνυμα που θα περάσουν στην Κομισιόν. Χαίρομαι που είμαστε εδώ, ε, χαίρομαι που έχουμε τους καλεσμένους που έχουμε από τους οποίους περιμένουμε να ακούσουμε συστάσεις και απόψεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε αμέσως δίνοντας άμεσα το λόγο στην Υπουργό κυρία ε, Μίντς. Λίδια Μίντς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Συμπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που αναλάβατε την πρωτοβουλία αυτής της συνεδριάσεως που μου επιτρέπει να ξαναθέσω στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας ένα φάκελο που αξίζει το ενδιαφέρον μας, όπως πολύ καλά το αναφέρατε. Η αντιπροσώπευση των γυναικών στα διηγητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Ζήτησα να συμμετάσχω ε, σήμερα στην συνεδρίασή σας και σε αυτή την ανταλλαγή ε, απόψεων έτσι ώστε να σας διαβεβαιώσω για την δέσμευση της ε, Λουξιβουριανής Προεδρίας να προωθήσει το φάκελο αυτό αλλά και γιατί εγώ προσωπικά του αποδίδω μεγάλη σημασία αυτού του θέματος. Γνωρίζετε ότι το θέμα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και ότι ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Είχα ήδη αναφερθεί σε αυτό που ε, πρέπει ακόμα να γίνει ε, την 14η Ιουλίου ενώπιον της Επιτροπής Γυναικών, όπου είχα αναφέρει ότι η ανισότητα ανδρών και γυναικών είναι μεγάλη στις θέσεις λήψης αποφάσεων και επομένως δεσμεύεται ε, η Λουξεμβουριανή Προεδρία στο πρόγραμμα εργασίας της να αναφερθεί στην ανάγκη ε, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αυτές τις θέσεις λήψης αποφάσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες έγιναν πολλά. Ε, εν είδη παραδείγματος θα ε, σας ε, μιλήσω για μια διεθνούς επίπεδου διάσκεψη 15 και 16 Οκτωβρίου στο Μοντόρφ Λεμπάν με το θέμα αυτό. Είχαμε μάλιστα παρουσία και της εισηγητρίας κυρίας ε, ε, Ρέγνερ, ε, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσία της εκεί, αλλά και για την πολύ θαραλέα της τοποθέτηση. Αυτό μας ε, επέτρεψε να έχουμε μία συζήτηση ε, υψηλού επίπεδου επί της ε, οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και πραγματικά αποτέλεσε εμβληματικό στοιχείο των συζητήσεών μας γιατί εκεί καταφέραμε να ε, βάλουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι εκπροσώπους του επιστημονικού, ακαδημαϊκού, οικονομικού και επιχειρηματικού κόσμου. Ε, εγώ μετά από τις δύο ημέρες τη διασκέψεως στο Μοντόρ Φλεμπέν κατέληξα και εγώ προσωπικά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο μέτρων έτσι ώστε να επιτύχουμε την επιθυμητή ε, η ισόρροπη ε, εκπροσώπηση των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια και σε θέσεις λήψης απόφασης. Δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις έτσι ώστε από τη μία στιγμή στην άλλη, ή από τη μία χρονιά στην άλλη να επιτύχουμε αυτήν την ισότιμη εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι ούτε πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένα καθολικό ε, φάρμακο για όλα τα προβλήματα. Ούτε αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελέσει ε, το θαυματουργό φάρμακο. Δεν είναι πανάκια, αλλά βοήθησε την κατάσταση σε πολλές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να εντάξουμε το κείμενο αυτό σε ένα γενικότερο πακέτο δεσμευτικών μέτρων που μπορεί να μας επιτρέψουν να προωθήσουμε τα πράγματα και μέσω των οποίων ε, μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. γιατί ε, μια νομοθετική βάση μπορεί να ε, ε, αποτελέσει ισχυρή βάση έτσι ώστε να δούμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Εγώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι δέσμοι μέτρων δεν θα είναι πλήρης, αυτό το πακέτο δεν θα είναι πλήρες εάν δεν συμπεριληφθούν και οι ποσοστώσεις. Και θέλω να το αποσαφηνίσω και ενώπιόν σας. Με το πνεύμα αυτό λοιπόν προετοιμάσαμε τα συμπεράσματα ε, σχετικά με, τις, ε, ε, με τη θέση όσον αφορά τη θέση των γυναικών που θα, στα συμβούλια, θέση που θα κληθεί να μελετήσει το Συμβούλιο Εύσκο της 7 Δεκεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε, διαπιστώνετε ότι το θέμα αυτό προχωράει με μάλλον θετικό τρόπο, μάλλον θετικό. Ε, είμαι ε, υπερήφανη γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία προχωρούν και προωθούνται, αλλά υπάρχουν και διάφορα ζητήματα τα οποία δεν προχωρούν με το ρυθμό που θα ήθελα. Υπάρχουν θέματα τα οποία Ε, απαιτούν πιο συλλογική ε, προσπάθεια και πιο ορατή δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών. Ε, το δε θέμα των γυναικών και τη θέση τους στα διοικητικά συμβούλια θα το αναφέρω σαν ένα θέμα που θέλει ακόμα μία όθηση από τους εμπλεκόμενους φορείς. Είχα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις 14 Ιουλίου και είχα υποσχεθεί ότι η Προεδρία ε, θα, είχε, έβαζε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Συμβουλίου. Ε, και επομένως ε, υποβάλαμε ένα συμβιβαστικό κείμενο. Ήταν απαραίτητο να υποβάλουμε ένα συμβιβαστικό κείμενο. και το κείμενο αυτό στην ουσία ήθελε να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς που είχαν εκφράσει τα κράτη-μέλη, τα οποία ήδη διαθέτουν εθνική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στις διάφορες αντιπροσωπείες τον απαραίτητο χρόνο να ε, μελετήσουν τις ε, προτινόμενες θέσεις. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία πρότεινε να αποσυρθεί το σημείο ε, από το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ της 5ης Οκτωβρίου. Ήταν απαραίτητο να αποσύρουμε λοιπόν το θέμα από την ημερήσια της 5ης Οκτωβρίου έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλες τις χώρες να μελετήσουν το θέμα έτσι ώστε να μην ε, μας κατηγορήσουν οι διάφορες κατηγορίες ή οι, ε, οι διάφορες εθνικές αντιπροσωπείες ότι ε, δεν, θα, ότι δεν είχαν την ευκαιρία ας πούμε να μελετήσουν ή να οικειοποιηθούν το περιεχόμενο του θέμ, εγγράφου αυτού και επομένως θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο επόμενο Συμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου ε, εν όψη γενικής ε, σύστασης. Αυτό θα ήθελα εγώ. Βεβαίως εμείς παραμένουμε ε, προσδεδεμένοι στις αρχικές φιλοδοξίες και στις πρώτες μας αρχές, ενώ ταυτοχρόνως παρέχουμε στις χώρες μέλη την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να συντονίσουν τις αρχές αυτές με τις εθνικές τους νομοθεσίες. Θεωρούμε ότι μια τέτοια ε, ευελιξία είναι απαραίτητη έτσι ώστε ε, να γίνουν σεβαστές οι εθνικές διαδικασίες οι οποίες είχαν θετική εξέλιξη σε ε, πολλές χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα σε, τεχνική, σε τεχνικό επίπεδο συζητιέται ακόμα. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι πραγματικά η στήριξη από τους πολιτικούς και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις εβδομάδες που απομένουν. Τις ε, προηγούμενες εβδομάδες ε, και μήνες προσπάθησα πάρα πολύ να πείσω τους Ευρωπαίους ομολόγους μου να αντιληφθούν τη συμβολική σημασία αυτή της πρότασης οδηγίας. Στους περισσότερους δεν χρειαζόταν να το πω γιατί όλοι αντιλαμβάνονται την ε, συμβολική σημασία. Τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα το γνωρίζουμε. Η Μία πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ της ε, πρότασης αυτής ε, θα ήταν ε, κατά την άποψή μου όχι μόνο ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις αλλά ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα για την ισότητα στην Ευρώπη. Αυτό μας χρειάζεται. Γι' αυτό το Συμβούλιο στις 17 ε, Δεκεμβρίου θα ασχοληθεί και με το μέλλον ε, της πρότασης οδηγίας και θα είναι, αποτελε... θα είναι με συγχωρείτε αποφασιστικός ο ρόλος του. Μπορώ να σας προσχεθώ πως η Προεδρία μας σε στενή συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια τις επόμενες εβδομάδες ε, και μήνες για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Νομίζω πως γνωρίζετε πως ε, πρόσφατος ε, στις αρχές της εβδομάδας μαζί με την Επίτροπο την κυρία Γιούνοβα συνέταξα μια επιστολή που απευθυνόταν σε όλα τα κράτη-μέλη για να τονίσω ξανά την ε, σημασία της πρότασης αυτής και να πω πως ε, είναι απολύτως αναγκαία για να καταπολεμήσουμε την ε, καταφανή υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οπότε αυτή τη στιγμή, τις επόμενες εβδομάδες, χρειάζεται να συνταχθούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή ε, ο σημαντικότερος σύμμαχός μου είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και το αντιλήφθηκα αυτό από τον Ιούλιο ήδη όταν παρουσίασα το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Για το ξεκάθαρο αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας της ε, πρότασής μας ήδη από το Νοέμβριο του 2013 αλλά και τις άλλες ε, πρωτοβουλίες τη σημερινή παραδείγματος χάρη να συνεδριάσουν από κοινού οι δύο επιτροπές αλλά και για τις πολλές και διάφορες συνεδριάσεις που εν μέρει δεν ήταν δημόσιες αλλά έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και βοήθησαν στις συζητήσεις με εθνικές κυβερνήσεις ή κοινοβούλια για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή και να βρούμε συμμάχους για την κοινή μας ε, υπόθεση. Οπότε θα τελειώσω εδώ την ε, παρέμβασή μου με μια περαιτέρω έκκληση να μην χαλαρώσουμε και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα τις επικριτικές φωνές που υπάρχουν ακόμα Υπάρχουν ακόμα κάποιοι που επικρίνουν, πρέπει να τους πείσουμε. για να βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες ε, να βρεθούν στα κέντρα αποφάσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ και για την στήριξη που μου δείξατε εξ αρχής και για την προσοχή σας σήμερα. Thank you, Lydia, for this Εγώ σας ευχαριστώ, Λίδια. Πάρα πολύ ευχαριστώ σαραλέα, αλλά τόσο ενθαρρυντική τοποθέτηση και πολύ στρατευμένη. Θα και την κυρία Ζωντάν από τον ε, Όσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλο προνόμιο ευκαιρία που έχω να συμμεριστώ μαζί σας στις εργασίες του ΩΣΑ για αυτά τα θέματα, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δεν θα σας εκπλήξει ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα και για το Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ και για τις 34 χώρες μέλη. Αρχικά θα ήθελα να σας ε, δώσω μια επισκόπηση σύντομα των συστάσεων του ΩΣΑ. some... Για αυτά τα πράγματα, ε, μερικά στοιχεία επίση και θα μοιραστώ και μερικές ιδέες που έχουμε για τα επόμενα βήματα. We do have... Λοιπόν, από το 2013 έχουμε εκδώσει συστάσεις για το φύλλο του όσα είναι ένα οριζόντιο πρόγραμμα συνολικό, καθολικό, δεν ξέρω πώς θα το λέγατε καλύπτει τρεις βασικούς τομείς την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Το θέμα των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εντάσσεται στο κεφάλαιο της απασχόλησης των συστάσεων. Όταν έχουμε μια σύσταση του Συμβουλίου, τόσα μέσα σε μια τριετία επανέρχεται το θέμα σε υπουργικό επίπεδο και γίνεται μια έκθεση ε, για το πώς ε, βαίνει η εφαρμογή. Έχουμε μια συνεχή αξιολόγηση δηλαδή και παρακολούθηση και αυτό θα γίνει ε, και θα υποβληθεί στους υπουργούς το 2017. Πολύ σύντομα. Οι συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο λοιπόν το ΕΣΑ για τις γυναίκες σε θέση λήψης ε, αποφάσεως, ιδιαίτερα σε διοικητικά συμβούλια, θέτουν πολλά ζητήματα. Τα δύο έχουν να κάνουν με την παρουσία του σε διοικητικά συμβούλια, ε, ποσοστώσεις, ε, θελοντικοί στόχοι, δημοσίευση και άλλα θελοντικά θέματα και πρωτοβουλίες. Εδώ λοιπόν βλέπετε το σύνολο των συστάσεων. Αυτό τι σημαίνει. Έχουμε και επιτροπές ε, στον ΩΣΑ οι οποίες ασχολούνται φυσικά ε, με τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Ε, σε αυτή την επιτροπή συμμετέχω και εγώ εκεί για την διοίκηση επιχειρήσεων. Όταν ενημερώνουμε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να συμπεριλαμβάνουμε και τις συστάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μας. Και G20 ε, ε, είχαν κάποιες συστάσεις που πρόσφατα αναθεωρήθηκαν και έχουν ε, δημοσιευθεί φέτος το φθινόπωρο. Και για πρώτη φορά τώρα συμπεριλαμβάνεται και αναφορά στις συστάσεις αυτές που δώσαμε για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβολία. Και τι λέγουν λοιπόν αυτές τις συστάσεις. Ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να πάρουν διάφορα μέτρα, ε, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στις δικές μας συστάσεις, για να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την ε, ποικιλία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και στις ηγετικέ ε, θέσεις των εταιριών. Ίσως κάτι που να είναι καινούριο για σας. Όταν συζητούμε για τα διοικητικά συμβούλια και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Αυτό έχει να κάνει και με τη σχέση μεταξύ των μετόχων, των διοικητικών συμβουλίων και της διοίκησης τη επιχείρηση. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί και εμεί το εντάσσουμε την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων όταν μετρούμε τις επιδόσεις, ε, τα προσόντα και ε, το έργο γενικά των διοικητικών συμβουλίων. Και όταν μιλούμε για γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, αυτό δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, ούτε θεωρητικό. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Και οι μέτοχοι πρωταγωνιστούν εκεί, αλλά κυρίως το διοικητικό συμβούλιο φέρει την κύρια ευθύνη για τα διαδικαστικά συγκεκριμένα για το διορισμό των μελών στα διοικητικά συμβούλια και θέλουμε να είναι σεβαστές αυτές οι αρχές με διαφάνεια. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το γενικό προφίλ και το ατομικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρει και την ευθύνη να εντοπίζει τους υποψηφίους, να τους ανοιχνεύει. Και αυτό γίνεται με επιτροπές διορισμών. Πώς έχει συζήτηση τώρα από τη δική μας σκοπιά. Από τη σκοπιά δηλαδή της διοίκησης επιχειρήσεων. Τι καθεστώς έχουν αυτές ε, οι αρχές. Όλα αυτά είναι προδιαγραφές και πρότυπα ε, θελοντικά. De facto τα χρησιμοποιούν όλες οι χώρες του κόσμου και η Παγκόσμια Τράπεζα ε, όταν συζητά θέματα προτύπων, κωδικών και προδιαγραφών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που όλα αυτά τα έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη μας και τα κράτη του G20 για να βελτιώνεται η παρουσία και η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Share with you, um, some of the research uh, and evidence. Να σας πω ποια είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά μας. Όλες οι συστάσεις βεβαίω που εκδίδουμε βασίζονται σε στοιχεία. Το 2012 πριν εκδώσουμε λοιπόν τις συστάσεις μας που έγινε το 2013, διαπιστώσαμε ότι όταν συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, ε, μπορεί να βελτιώνει τη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν πολύ κακές επιδόσεις. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει κάπως να το συγκεκριμενοποιήσω. Σήμερα βεβαίως έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι πριν από τρία χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέση και θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια μεταξύ διαφόρων στοιχείων. Είναι πολύ δύσκολο ε, να αποδείξουμε ότι υπάρχει ε, σχέση αιτίου και αιτιατού. Στην έκθεση του 2012 λοιπόν θέλω να σας αναφέρω μερικά στοιχεία που θα αναθεωρηθούν. Όταν έχουμε ένα ετερογενές διοικητικό συμβούλιο αυτό είναι θετικό. Ε, υπάρχουν τα περίφημα δίκτυα των old boys που δεν συμμετέχουν πάρα πολλές γυναίκες και δεν λαμβάνονται πάντα αποφάσεις στα διοικητικά συμβούλια. Επίσης, είναι Φυσικά πιο πλούσια τα διοικητικά συμβούλια όταν έχουν συμμετοχή γυναικών με διαφορετικές ε, απόψεις και τρόπους επίλυσης διαφόρων ζητημάτων. Εμπλουτίζεται λοιπόν ε, η δίκη των επιχειρήσεων από την παρουσία των γυναικών. Ε, αυτά τα έχουμε μετρήσει, είναι στοιχεία που έχουμε δει. Τώρα, ε, στις δικές σας ιστοσελίδες έχουμε δει ότι 20,2% ε, στις μεγάλες εταιρείες ε, καλύπτονται από γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και μόλις 3,3% είναι εκτελεστικοί διευθυντές, CEOs, γυναίκες, διευθύντριες δηλαδή. Αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και θα πρέπει να το τονίσουμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ενώ είναι 20% οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, είναι μόνο 3,3% εκτελεστικοί διευθυντέ. Εννέα χώρες μόνο έχουν ε, περάσει το όριο του 20% των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι μια έρευνα ε, που έγινε το 2014 και στις ε, κορυφές είναι πολύ μικρή η αλλαγή, το 3,3% παραμένει από το 2014. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας και δεν θέλω να επεκταθώ ή να ε, βαθύνω πάρα πολύ σε αυτό, αλλά στις οικονομικές επιδόσεις, στην απόδοση των μετοχών και προφόρο, στα προφόρων έσοδα, αυτά αυξάνονται όταν είναι περισσότερες οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και τις εκτελεστικές επιτροπές. With uh, more women on boards, ten... Οι εταιρείε που έχουν περισσότερε γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια έχουν και λιγότερε συγκρούσει. Ε, στη διακυβέρνηση και στη διοίκησή τους. Γι' αυτό το μετρήσαμε. Και μπορείτε να το διαπιστώσετε σε 6.500 διοικητικά συμβούλια μειώνεται κατά πολύ ο κίνδυνος όταν συμμετέχουν γυναίκες Σας είπα ότι υπάρχουν διάφοροι πρωταγωνιστές, αν τώρα στους μετόχους και αυτοί δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες. Όπως σας είπα είναι και καλύτερε επιδόσεις, οπότε κατάλαβαν και οι επενδυτές ότι έχουν συμφέρον να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 τρεις μεγάλοι επενδυτές είπαν ότι θα αρχίσουν ε, να ε, απορρίπτουν στις αιτήσει γενικές συνελεύσεις τους 250 εταιρείες που έχουν αμυγός ε, ε, ανδρικό διοικητικό συμβούλιο 100%. 126 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Καλιφόρνια το 2014 δεν είχαν καθόλου γυναίκες στα διοικητικά του συμβούλια. Και είναι ακόμα πάρα πολλά τα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας αναφέρω. Ε, μια άλλη ενδιαφέρουσα στατιστική που μόλις είδα από μια φετινή μεγάλη μελέτη και πάλι και έρευνα ε, του Bordex είναι το κόστος που συνδέεται ε, με τα αμυγός ανδρικά διοικητικά συμβούλια. Σε 1050 εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ινδία ε, διαπιστώθηκε ότι χάνουν ευκαιρίες της τάξεως των 655 δισεκατομμυρίων σε αυτές τις χώρες εταιρείε που δεν έχουν καθόλου γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. This is just a quick snapshot. Αυτά λοιπόν λέει ο ΣΑ είναι ένα στεγμιότυπο μόνο φωτογραφικά σας λέω ότι συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που έχουν ε, υποχρεωτικέ ποσοστώσεις και τις έχουμε μελετήσει και αυτές. Άλλες που χρησιμοποιούν πιο, ήπι, πιο ήπιες μεθόδους με θελοντική συμμετοχή, με όχι δεσμευτικούς στόχους. Θα κάνουμε λοιπόν μια έκθεση προόδου και με μεγάλη χαρά να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και πώς συνεχίζετε το έργο σας προς την κατεύθυνση αυτή. Στην έκθεσή μας λοιπόν θα δούμε ποια ήταν η επίπτωση των διαφόρων προσεγγίσεων και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία. Ε, όταν υπάρχει αυτή η επιτυχία για ποιο λόγο συμβαίνει, πού οφείλεται και υπάρχουν και συστάσεις του G20 και του ΩΣΑ για τις γυναίκες, τις επιχειρήσεις Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιοποιείται το ταλέντο και οι δεξιότητες όλου του πληθυσμού, γιατί αλλιώς χάνουμε ευκαιρίες. Και επίση να δούμε ποιες είναι οι διάφορες δυνάμεις, μέθοδοι που αλλάζουν τις νοοτροπίες, τις πρακτικές και βελτιώνουν την κατάσταση. Ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε κάθε φορά να εξαγάγουμε. Αυτά Ευχαριστώ πολύ. Mm, thank you very much for this very interest. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Μετά την ε, ίσως πιο απεσιόδοξη νότα προηγουμένως, μας δίνει κάποιες ελπίδες. Αρχίζει η συζήτηση λοιπόν προτείνω. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις. Η Μαρή Αρένα. Euh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις ε, παρουσιάσεις. Δυστυχώς ε, ε, ήμουν σε άλλη πολύ σημαντική συνεδρίαση για τα για τα δικαστήρια, τα διαιτητικά δικαστήρια και το ISDS και δεν ήμουν από την αρχή εδώ. Εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι γιατί δεν καταφέρνουμε επιτέλους να πείσουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει όσον αφορά το θέμα αυτό που αφορά την βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια. Η πρόταση είχε γίνει από την Κομισιόν και την, ε, προ... στήριξε και το Κοινοβούλιο και είναι μια πρόταση η οποία βεβαίως είναι φιλόδοξη αλλά δεν είναι εξαιρετικά δεσμευτική όσον αφορά τις κυρώσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Πιστεύω ότι ε, το, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας σήμερα επιτρέπει στις χώρες που έχουν την βούληση αυτή να προχωρήσουν πιο γρήγορα όσον αφορά την ισομερή εκπροσώπηση. Δεν αφορά μόνο φεμινιστικά ε, επιχειρήματα αλλά και οικονομικά γιατί φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει αυτή η ποικιλία εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια πέρα από το ε, φεμινιστικό καθαρά επιχείρημα που θα μπορούσε να είναι το δικό μου επιχείρημα υπάρχουν και τα οικονομικά επιχειρήματα και εξάλλου όπως είπα και προηγουμένως δίνει τη δυνατότητα το κείμενο αυτό, η πρόταση αυτή στα, ε, ε, στις χώρες μέλη να προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό. Θα θέλαμε λοιπόν να με τη βοήθεια και της κυρίας Υπουργού να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς στο Συμβούλιο, να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση και γιατί δεν, προωθεί, ε, δεν προωθείται η συζήτηση δηλαδή ήθελα μια πολιτική ερώτηση για το τι συμβαίνει ακριβώς στο μυαλό του Συμβουλίου. Πρόεδρος, ωραία, να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις και να, απαντήσει, να απαντήσουν οι δύο κυρίες από κοινού. Ναι, κύριε Πεθέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, για τη συντομία σας και για την αποφασιστικότητά σας και τις δύο και την κυρία Μούς και την κυρία ε, Τζούρνταν. Ήταν πάρα πολύ εύλογα όλα αυτά που μας είπατε και πάρα πολύ κατατοπιστικά. Περιγράψατε την κατάσταση. Ε, είναι τόσο βαρύ, το, το, τόσο μεγάλο το βάρος δηλαδή της κατάστασης, της αλήθειας, της περιγραφής, οπότε τι τρέχει, πούμε, γιατί δεν προχωράει η κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι, είναι συντριπτική και το μόνο που στον κόσμο είναι ίσα μοιρασμένο είναι το φύλλο, το ταλέντο, οι δεξιότητες και οι ικανότητες. Όλα τα άλλα όταν δεν αξιοποιούνται πάνε χαμένα. Λοιπόν αυτό τι είναι τώρα σπατάλη, αδικία και τα δύο κρίμα δεν είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω και την ε, κυρία Υπουργό για τα επόμενα βήματα γιατί Μιλήσατε για την ε, προσοχή έγκριση ε, στο Συμβούλιο και για την ε, αναστέλουσα μειοψηφία. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως εκεί, γιατί ξέρουμε και η επόμενη Προεδρία είναι η Ολλανδία και ξέρουμε και ποια είναι η στάση της. Οπότε τι θα κάνουμε εκεί. Η μία Προεδρία θα διαδέχεται την άλλη και θα το μεταβιβάζει το θέμα στο διάδοχό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Λέει κανονικά θα έπρεπε να εγκριθεί το 16. Αυτό είναι ευσεβής πόθος, είναι εντολή, είναι απόφαση. Ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέση της. Διότι ούτε η ίδια δεν κατάφερε να το επιβάλλει ε, τη στιγμή που συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτό ήταν στα χέρια τους και είναι κρίμα και πάλι. Όπως και από τις εταιρείε εμείς ζητούμε να παρακολουθούν, να είναι με διαφάνεια επιλογή και ο διορισμός των γυναικών και των εκπροσώπων, θέλουμε κι εμείς να δικαιολογείται αυτό, να μην υπάρχει λοιπόν καμία ε, υποψήφια που να ε, είναι σε θέση να αναλάβει μια θέση με αξιοκρατικά κριτήρια και να μην λαμβάνεται αυτό υπόψη. Και θα πρέπει τα ίδια κριτήρια που ζητάμε από τους άλλους να τα επιβάλλουμε και στον εαυτό μας και να έχουμε και μακροπρόθεσμους ε, στόχους που είναι το, η Ατζέντα 2030 ε, των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί συμμετέχουν και όλα τα μέλη μας. Και ο πέμπτος στόχος είναι ισότης. Αυτά δεν είναι ε, στόχοι που πρέπει να επιβάλλουν κάποιοι δωρητές κάποιους δικαιούχους οικονομικής αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό δεσμεύει όλα τα κράτη και όταν υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης οικονομικής μεγέθυνσης ή, όταν υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη του ανθρώπου, α πούμε, όταν κάποιο παιδί βλέπουμε τα δόντια του να βγαίνουν στραβά, του βάζουν σιδεράκια και του τα διορθώνουν, δεν του, δεν του τα αφαιρούν. Λοιπόν, είπαμε ποια είναι η πραγματικότητα, αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται και στη διοίκηση των επιχειρήσεων όταν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν εμπειρογνώμονα, γιατί πρέπει να είναι ένα εμπειρογνώμο, δεν μπορεί να είναι και μία εμπειρογνώμο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ε, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα αυτή η κατάσταση που ζούμε. Και αν χρειάζεται κάποια διόρθωση, το 2018-2020, ξέρω εγώ, να διορθώσουμε την κατάσταση. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα έχουμε ένα προσδόκιμο ζωής γύρω στα 80 έτσι. Έτσι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα χάσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο ή θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε και τις πρόοδες που κάνουν τα διάφορα κράτη. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Marino Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ και την κυρία Ζωνταν και την ε, κυρία Υπουργό. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο, μια κοινή συνεδρίαση δύο επιτροπών και πραγματικά ε, λείπουν πολλοί βουλευτές και δεν είναι σωστό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για να μην είμαστε όλοι παρόντες. Να σας πω κάτι κυρία Υπουργέ. Κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να με κάνει υπερήφανο. Για πολλά χρόνια ήμουν πρόεδρος ε, της, ε, ε, της Ένωσης Δικηγόρων της Πορτογαλίας για δύο θητείες μάλιστα του Δικηγορικού Συλλόγου της Πορτογαλίας για δύο συνεχόμενες θητείες. Αυτό έγινε βέβαια πριν από αρκετά χρόνια. Όταν έφτασα, όταν έγινα πρώτη φορά πρόεδρος του Διακορικού Συλλόγου, ε, στην, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, υπήρχαν μόνο τρεις γυναίκες. Εγώ όμως ε, ήθελα να αλλάξω την κατάσταση αυτή. Ε, όμως στάθηκε πάρα πολύ δύσκολο να βρω γυναίκες ε, έτοιμες να πάρουν την ε, θέση αυτή. Γιατί στην ε, Πορτογαλία μπορεί να είναι μια γυναίκα δικηγόρος, αλλά είναι ταυτόχρονα και σύζυγος και μητέρα και έχει ένα σωρό άλλα πράγματα στο κεφάλι της και έγνοιες με, μετά από ε, μεγάλη προσπάθεια κατάφερα ε, να βρω τις γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να δεχτούν τη θέση αυτή και εν τέλει αποτέλεσαν μεγάλο πλούτο για το δικηγορικό σύλλογο. Όταν έφυγα υποστήριξα την ε, υποψηφιότητα μιας γυναίκας ε, ε, στο, σαν ε, υποψήφιας προέδρου του δικηγορικού ε, συλλόγου. Και μάλιστα ο σύλλογος μας πλέον είχε στο διοικητικό του συμβούλιο πλειοψηφία γυναικών. πραγματικά αυτό με έκανε πάρα πολύ περήφανο. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Πορτογαλία γιατί παραδοσιακά ε, το δικηγορικό επάγγελμα ε, έχει σαφώς περισσότερες, περισσότερους άνδρες από ότι γυναίκες. Θεωρείται ανδρικό επάγγελμα. Ακόμα πολύ πρόσφατα αναφέρθηκα σε μία παρέμβασή μου ε, ενώπιον του ε, δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπέρ των γυναικών δικαστών. Και τώρα αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εμείς να ζητούμε στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων να έχουν γυναίκες μέλη, ενώ εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σεβόμαστε αυτήν την αρχή της ισοτιμίας και της ίσης αντιπροσώπευσης. Και ε, μάλιστα αυτό που το επιχείρημα το οποίο ακούμε όταν υποβάλλουμε ένα τέτοιο ερώτημα είναι ότι ε, δεν ε, μας το επιτρέπει το, ε, η συνθήκη λειτουργίας αλλά αυτό ε, είναι πάρα πολύ σοβαρό και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί εμείς μιλάμε εδώ για τις επιχειρήσεις, μιλάμε για τις ε, ε, υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις, αλλά εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν σεβόμαστε αυτές τις αποφάσεις. Οι γυναίκες δεν έχουν ίδιες ευκαιρίες. και ακριβώς γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει οι γυναίκες να μην έχουν, ε, ε, να είναι ελεύθερες και να μπορούν να κανονίσουν τη ζωή τους, να ρυθμίσουν και να οργανώσουν τη ζωή τους όπως θέλουν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε στις χώρες μας να υπάρχουν ακόμα ε, εγκλήματα κατά των γυναικών, βιαιότητες οι οποίες ε, ε, έχουν σαν μόνο υπόβαθρο το φύλλο της γυναίκας. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον καταστάσεις οικογενειακής βίας, βίας κατά των γυναικών, γιατί εγώ βλέπω, παίρνω παράδειγμα από τη χώρα μου που το πρόβλημα αυτό είναι τραγικό. Έχει πάρει τρομερές διαστάσεις. Ευχαριστώ πολύ ε, που είσαστε εδώ ε, και ε, βεβαίως λέω ότι καλό είναι να ασχοληθούμε με τα διοικητικά συμβούλια αλλά να ασχοληθούμε και με την κατάσταση και πιο χαμηλά. Πρόεδρος. Αδελφοί, μία ώρα είχαμε οπότε παρακαλώ οι επόμενοι μιλητές να είναι κάπως πιο σύντομοι στις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πρώτα. Θέλω να ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτή και να ζητήσω συγγνώμη. Διότι παράλληλε υποχρεώσει δεν μα επέτρεψαν να είμαστε εδώ από την αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Μούτ και να ζητήσω και εγώ κάτι που ζήτησαν οι συνάδελφοι δώστε μια τελική όθηση σε αυτή τη πρωτοβουλία, να προχωρήσει τουλάχιστον ένα βήμα στα θέματα της ισότητας. Βεβαίως δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που μας απασχολεί και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα αρχίζουν να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και το μέγα πρόβλημα είναι ότι ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες, εδώ και αρκετό χρόνο πλέον, έχουμε νομοθεσία και βέλτιστες πρακτικές που είναι πολύ πιο προ και χωρημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικός μας ρόλος λοιπόν θα πρέπει να είναι να είμαστε ε, ηγετική δύναμη σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχουν ξεπεράσει τα κράτη και οι περιφέρειες. Και οι γυναίκες να καταλαβαίνουν ότι είναι Ευρωπαίες ε, και να ταυτίζονται με αυτό. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τι να την κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αν οι περιφέρειες και τα κράτη έχουν πιο προηγμένη νομοθεσία. Επίσης, έχουμε ανησυχητικά στοιχεία για την έμφυλη βία. Αλλά και κάτι άλλο που μας θορύβησε πάρα πολύ. Το είπαν οι συναδέλφοι σας, γιατί το συζητήσαμε με την πρόεδρο της Επιτροπής μας ε, και με την Επιτροπό και με την κυρία Μπεσέρα. Και ακούμε ότι τα θέματα της ισότητας και οι πρωτοβουλίες για την κακομεταχείριση στην Ολομέλεια μπαίνουν πάντα τελευταία ώρα, νυχτιάτικα, και είμαστε πέντε γυναίκες που συζητάμε άγρια μεσάνυχτα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, αυτό το καθημερινό, πώς να το πω, ψωμοτήρι και αυτό που δείχνουμε προς τα έξω είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα θέματα των γυναικών γιατί τα βάζουμε τελευταία ώρα τη νύχτα. Ευχαριστώ λοιπόν και την κυρία Ζούρταν και θέλω να την ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε για την εμπειρία που έχετε με τις ποσοστώσεις, ότι είναι, λέτε, ε, μια εφελούσια ρύθμιση αυτή. Και παρόλα αυτά έχετε διαπιστώσει ότι έχουν κάποια σχετική επιτυχία. Εκείνες οι εταιρείες που έχουν γυναίκες στα διοικητικά του συμβούλια, τι κίνητρα είχαν, μόνο οικονομικά ή υπήρχαν και άλλα ελαττήρια, ξέρω εγώ, ε, θέματα ευελιξίας του ωραρίου, συμφιλίωσης του ε, οικογενειακού με τον εργασιακό βίο. Για ποιο λόγο, αφού είναι θελοντικό αυτό το σύστημα και όχι υποχρεωτικό, επέλεξαν οι εταιρείε να βάλουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκούτλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το πάνελ. Σα ευχαριστώ και σας κυρία Μούτς, κυρία Υπουργέ, για στο που μας είπατε. Αλλά μου έδωσαν ελπίδα. Αλλά αναφέρατε και τι αντίσταση συναντάμε και εκεί πέρα ανησύχησα. Επίσης, Ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας για τον ΩΣΑ. Και βεβαίω πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την απόψή σας για το ποιο οικονομικό όφελος θα μπορούσαμε να δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν προχωρούσαμε με μια καλύτερη ισορροπία όσον αφορά το θέμα αυτό στα διοικητικά συμβούλια. Γιατί θα ήθελα να πω πως θεωρώ πως βλέπω πως ε, ε, το να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες θα έχει θετικό αποτέλεσμα, θα έχουμε πρότυπα και όλες οι γυναίκες ε, που μορφώνονται και θα αποκτούν τα προσόντα αυτά θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες. Είναι λοιπόν θέμα δικαιωμάτων και ίσου ανταγωνισμού. Στην Σουηδία, παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες ε, είναι πιο εκπαιδευμένες από τους άντρες αλλά έχουμε μια ευκαιρία εδώ πέρα οικονομική ευκαιρία και θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις εταιρείε μας στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για το τι είδους οικονομικό όφελος θα έχουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα όταν θα το συζητήσει το θέμα το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κυρία Μασκά. Ευχαριστώ σύντομα γιατί το ήθελα και εγώ να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε η κυρία Μαρία Ρένα κάπως πιο λεπτομερό στο ερώτημα είναι το εξής πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πείσουμε αυτούς που είναι κατά μιας τέτοια ευρωπαϊκής οδηγίας. Ε, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πρακτικά πλέον αποτελέσματα που λένε ποια είναι τα ωφέλη από κάτι τέτοιο με μια οδηγία με την οποία όλοι συμφωνούν ότι είναι φιλόδοξη αλλά όχι τόσο καταναγκαστική. Στην ε, Ιταλία είχαμε μία σειρά συζητήσεων πάρα πολύ έντονων για αυτό το θέμα παρά το ότι εμάς η νομοθεσία μας ήταν πολύ πιο επιτακτική. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ Μάρκ Ταραμπέλα. Να συνεχίσω κι εγώ την ίδια σκεπτική. Η κυρία Ζουρντό του ΩΣΑ μας έδειξε, μας είπε ότι υπάρχουν σαφή οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία θα απορρεύσουν από την ισοτιμία ε, του ανδρών και γυναικών. Η κρίση του 2008 ε, ε, απέδειξε ότι οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες των οποίων τα διοικητικά συμβούλια είχαν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αντιστάθηκαν καλύτερα στην κρίση. Ε, ο Γκάμπριελ Σένα και ο συντηρητικός και ενάντια στην ε, θέση των φίλων του ε, πήρε κάποιες αποφάσεις προς την, κατεύθυνση αυτή και ενώ στην αρχή όλοι ήταν αντίθετοι τελικά έφτασε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τρίτο, είμαστε πολιτικοί, όχι διπλωμάτες. Εγώ σέβομαι απόλυτα τους, δημοκρα... τους διπλωμάτες αλλά δεν μιλούν με την ίδια ευθύτητα που μιλάμε εμείς και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Μόσκα προηγουμένως ε, ε, η Γερμανία έχει ας πούμε μια πιο ένα πιο δεσμευτικό κανόνα ε, και λέει τώρα «Α, εμείς δεν χρειαζόμαστε γιατί εμείς τα έχουμε κανονίσει στη χώρα μας». Μα αυτό είναι εγωισμός. ή όπως οι Σουηδοί οι οποίοι λένε «Εμείς δεν θέλουμε να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανόνας για τις μητρικές άδειε, γιατί εμείς ήδη το έχουμε ρυθμίσει το θέμα». Ναι, εντάξει υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να αλλάξουν γιατί είναι υπερσυντηρητικές κτλ κτλ. Άλλε οι οποίε δεν θέλουν να αλλάξουν γιατί ήδη έχουν αλλάξει προηγουμένω οι, οι ίδιες. Ε, θα δούμε τώρα ποια είναι η ανασχετική πλειοψηφία, ε, μειοψηφία συγγνώμη, στο Συμβούλιο. Αυτό δεν το ξέρω, πρέπει να δούμε ε, τι λένε οι συνθήκε. Επίση θα πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι και για ποιο λόγο μπλοκάρουν. Ε, ακούσαμε μόλι ότι οι κάτω χώρε, χώρα που θα σα διαδεχτεί στην Προεδρία κυρία Υπουργέ, μπλοκάρει. Αλλά νομίζω ότι οι κάτω χώρε είναι μια χώρα όπου πραγματικά τα δικαιώματα των γυναικών έχουν προστατευτεί περισσότερο από ότι άλλες, σε άλλες χώρες. Επομένως θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να καταλάβουμε ποιος μπλοκάρει τι και γιατί. Πολύ ωραία τα είπατε λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Λεγκρίπ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω, μια και παίρνω το λόγο μετά από πολλούς άλλους ομιλητές, να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη αλλά εγώ, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ε, ε, θα ήθελα ε, να ξέρω, να έχω πληροφορίες πιο συγκεκριμένες, γιατί έχουμε βέβαια κάποιες διαρροές, έχουμε κάποια άρθρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι πραγματικά οι χώρες, από εσά που τα ξέρετε από πρώτο χέρι, ποιες είναι οι χώρες που μπλοκάρουν την διαδικασία. Εγώ ε, προέρχομαι από τη Γαλλία, μια χώρα η οποία ε, πριν από 50 χρόνια κιόλας ε, σε μια περίοδο μάλιστα πλειοψηφία που θα μπορούσε να οριστεί ως συντηρητική έναν νόμο όσον σχετικό με τις ποσοστώσεις ε, ο οποίος νόμος είναι πολύ ε, ενδιαφέρον. Πολλά έχουμε πει όσον αφορά ε, το ενδεχόμενο κοινωνικό συγγνώμη, οικονομικό όφελος όσον αφορά την συμμετοχή των ε, γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, ε, πρέπει να σας πω ότι 28 δις δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο σε 10 χρόνια μπορεί να είναι ε, το, το όφελος του ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε μια πραγματική ισοτιμία ανδρών γυναικών στον, στους χώρους εργασίας. Αυτά ήθελα να σας πω και θα ήθελα να σας ζητήσω ζητήσω να απαντήσετε άμεσα στην ερώτηση που κάνουμε σχετικά με τις χώρες που μπλοκάρουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εσείς και η κυρία Γκάμπριελ, κοιτάξτε, μια που μίλησαν όλοι τόσο πολύ, θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Ζορντάν. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ο ΣΑ δεν ρωτάει γιατί χρειαζόμαστε τις γυναίκες στα Ρωσού, αλλά το πώς. Πλέον το ζήτημα είναι το πώς. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι η παρακολούθηση. Πώς αντιδρούν οι χώρες σε αυτή την παρακολούθηση όταν δεν σημειώνουν πρόοδο, πώς ε, θα μπορέσουμε να τις πείσουμε να πάρουν τα πράγματα κάπως πιο σοβαρά. Τα παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά με οικονομικά επιχειρήματα. Οπότε πείτε μας δύο-τρία λόγια ακόμα, όπως είπαμε, για την εποπτεία αυτή την παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις ε, άκουσα εγώ για την κυρία Ζουρντάν και περισσότερες ε, για την άλλη, για την κυρία Μούτσου. Ας ξεκινήσει λοιπόν η κυρία Ζουρντάν. Σας ευχαριστώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τις απόψεις ε, και τις ερωτήσεις σας για το θέμα της ε, ποσόστοσης. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα όπως με οποιοδήποτε άλλο μέτρο, κανονισμό, νόμο ή εθελοντική ρύθμιση, το θέμα που ρωτάμε πάντα ήταν ποιος ήταν ο αρχικός στόχος. Οπότε όταν κοιτάμε τις ποσοστώσεις ε, και τι αντίκτυπο έχουν, αυτό το ερώτημα θέμε να κάνουμε. Και αν δείτε κάποιες περιπτώσεις όπως η Νορβηγία, ναι, έχουν φτάσει τον στόχο του 40% στα δουσού, αλλά ο στόχος είναι γενικώ περισσότερες γυναίκες ε, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε εκτελεστικές επιτροπές ε, και επικεφαλής ε, εταιριών και δεν το έχουν πετύχει αυτό πλήρως. Αυτό ακριβώς κοιτάμε για να δούμε ποιε ποιες είναι οι σχέσεις και γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Και τι άλλο πρέπει να γίνει. Και επίσης συνεργάζομαι πολύ με Ασία και αν δείτε την Ινδία που μόλις έβαλε στον, στο εταιρικό δίκαιο το μήνυμο μίας γυναίκας αναδέλτα σίγμα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και μία αν έχουν μία γυναίκα θα είναι κάποια συγγενής ε, κάποιου. Μπορεί να έχει τα προσόντα, αλλά θα δείτε πολλές εισηγμένες εταιρείε ε, που θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το γράμμα του νόμου, αλλά δεν θα είναι ένα άτομο που θα έχει τα προσόντα. Θέλουμε αποτελεσματικά ΔΣ να ανοίξουν τις διαδικασίες επιλογής σε όλες τις υποψήφιες και οι υποψήφιες να είναι προετοιμασμένες να αναλάβουν αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Και δεν είναι μόνο ο νόμος που θα βοηθήσει να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Το θέμα λοιπόν για την παρακολούθηση είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Τι κάνουμε λοιπόν, έχουμε μια επιτροπή διοικητική όπως λέγεται με συμμετοχή 34 χωρών, θα τους αποστείλουμε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Ε, δεν βαθμολογούμε τις χώρες. Κάνουμε μια σύγκριση. Και ακόμα και χώρες όπως η Ιαπωνία, που είναι πολύ πίσω. Νομίζω η Κορέα και η Ιαπωνία είναι στον πάτο. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ γιατί με την ε, τωρινή κυβέρνηση υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά, της, στο πρόγραμμά τους ε, στην Ιαπωνία. Οπότε ακόμα και η Ιαπωνία το σκέφτεται σοβαρά και χρησιμοποιούν τον όσα για να στηρίξουν αυτούς που θέλουν να προχωρήσει το θέμα αυτό. Οπότε είμαι αισιόδοξη για τα αποτελέσματά μας. Βεβαίως πάντα εμείς κάνουμε την έρευνά μας δεν βασιζόμαστε μόνο στις απαντήσεις ε, των κρατών μελών, αλλά τελικά είναι μια καλή βάση για μια σωστή συζήτηση, αυτό το οποίο θα θέλαμε δηλαδή. Να δούμε. Πριν ε, δώσω τον λόγο στην Υπουργό, να ρωτήσω τον κύριο Στάιν από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη αν θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο για την οργάνωση της εκδήλωσης αλλά για την συνεχή του στήριξη για την οδηγία αυτή και να ευχαριστήσω και την Προεδρία του Λουξεμβούργου, την κυρία Υπουργό για την στενή συνεργασία και τις προσπάθειες που καταβάλουν και την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδουν σε αυτή την πρόταση. Όταν η Κομισιόν υπέβαλε αυτή την πρόταση πριν από τρία χρόνια γνώριζε ότι θα είναι κάτι το επίμαχο και υπάρχουν εδώ πέρα αποκλίνουσες απόψεις ε, μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς ορίσαμε ξεκάθαρους στόχους ε, και προθεσμίες αλλά δεν βάλαμε συγκεκριμένη ποσόστοση. Διαλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση και καταλήξαμε στην διαδικασία επιλογής για το ΔΣ και χαίρομαι που το ανέφερε και η βουλευτή σας. Και θεωρούμε πως η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές θα μας, πάει, μας προχωρήσει πολύ στην κατεύθυνση επίτευξης αυτών των στόχων. Τώρα, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει αυτή την προσέγγιση, δεν έχετε αλλάξει τη φιλοσοφία του κειμένου. Το έχετε εγκρίνει με κάποιες τροπολογίες και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που τώρα είναι σχεδόν στο τρίτο έτος στο Συμβούλιο η Κομισιόν με ένα τρόπο μετρούσε την πρόοδο και αυτό ήταν εάν το κείμενο παραμένει στο πνεύμα της ε, πρότασης. Δηλαδή να έχει δεσμευτικές ε, διατάξεις με ευελιξία για τα κρατη αλλά υπό έναν όρο ότι θα επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα. Οπότε παρακολουθήσαμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και μπορώ να πω πως το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο παραμένει πιστό στην φιλοσοφία της πρότασης. Γι' αυτό Έχουμε κάνει πολλή δουλειά εδώ πέρα με διάφορες προεδρίες. Εμείς θεωρούμε πως το κείμενο είναι όριμο για υιοθέτηση. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση της κυρίας Υπουργού πως θα είναι αποφασιστική η συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στις 7 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν και ο Επίτροπος να έχει ρίξει το πολιτικό του βάρος εδώ πέρα και προσπαθούμε ακριβώς να το προωθήσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα, είναι καθαρά πολιτικό. Να πείσουμε τα κράτη-μέλη δηλαδή που δεν έχουν πιστεί να στηρίξουν την πρόταση αυτή. Εμείς από την πλευρά μας, η Προεδρία από την δικιά της ε, και θέλουμε βέβαια στήριξη από βουλευτές ε, για να επηρεάσουν τις ε, κυβερνήσεις τους. Ε, πρόκειται για μια στιγμή κρίσιμη και θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε τώρα ακριβώς ε, να εμπλακείτε. Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ε, οι εξαιρετικές παρεμβάσεις της κυρίας Ροδόν και του κυρίου Στάινα ε, με οδηγούν στο να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα σας απογοητεύσω γιατί ε, δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι υπεύθυνοι για το μπλοκάρισμα. Δεν θα καταδώσω κανέναν. Άλλωστε οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ναι, προβληματίζομαι όντως, αλλά δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου εν ώψη της, ε, του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου, ε, όπως σας είχα πει ήδη από την αρχή, κρατώ τις ε, ελπίδες μου. Σας είχα πει κιόλας ότι είχα αποσύρει από τη μερίσια διάταξη του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου το θέμα αυτό, έτσι ώστε να επιτρέψω σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των διστακτικών χωρών, ε, να δώσω, λέω, την ευκαιρία σε όλες τις χώρες αυτές ε, να συζητήσουν αυτήν την πρόταση που δεν είναι πολύ δεσμευτική, δεν είναι υπερβολικά δεσμευτική, έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, είναι φιλόδοξη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσει. Βεβαίως έχουμε ακόμα το περιθώριο να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση για το θέμα αυτό. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι δεν είναι πολλοί οι βουλευτές ε, που είναι σήμερα παρόντες. Ε, εγώ ε, πραγματικά ευχαριστώ από καρδιά σε τους βουλευτές που παρίστανται, αλλά βλέπω ότι είναι αρκετοί ε, είναι πολλοί λοιπόν αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν και εξ και των ε, συναδέλφων, εξ ε, και χωρών που διστάζουν ακόμα για να τους δώσουν έτσι αυτή την όθηση που χρειάζονται να τους ενθαρρύνουν τους υπολείπους. Μα ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που μπλοκάρουν τώρα, μην με βάζετε να σας λέω τέτοια πράγματα. Η οδηγία αυτή, το είπατε και εσείς άλλωστε, έχει εμβληματικό χαρακτήρα. Μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ε, μήνυμα. Και ευγνωμόνω την κυρία Ζουρντόν γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για την κάλυψη ενός δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά γιατί βάσει πολλών μελετών ε, προκύπτει ε, με βεβαιότητα ότι ε, υπάρχει σαφής ε, ε, σχέση και με την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας και επομένως μιλάμε για μία απόφαση η οποία ε, θα ξεπεράσει όλες τις προκαταλήψεις οι οποίες εμποδίζουν τις γυναίκες να λαμβάνουν υψηλές θέσεις απόφασης με οικονομικό χαρακτήρα η βουλευτής από την Ισπανία το είπε ότι ούτως ή άλλως ποτέ δεν προχωρούν τα θέματα ισότητας με πολύ γοργό ρυθμό και συμφωνώ με τη διαπίστωση αυτή. Σημερίζομαι την άποψή σας ε, κύριε Βουλευτά και το είπε και ο κύριος Πίντο γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για τη θέση της γυναίκας μονάχα ε, στις, ε, στην οικονομική σφαίρα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για, την, ε, για τον νομικό κόσμο, για τον κόσμο της εργασίας γενικότερα κάθε φορά είναι διαφορετική η διαδικασία, αλλά η κατεύθυνση, ο στόχος είναι ίδιος. Όπως ε, σας είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει θαυματουργή λύση. Υπάρχουν πολλά μέτρα, πολλές δέσμες μέτρων ε, που ε, θα πρέπει να υλοποιηθούν είτε με δεσμευτικού χαρακτήρα είτε προαιρετικού. Και να σας πω ότι για μένα αυτή η δέσμη, το είπα και από την αρχή, δεν μπορεί να είναι πλήρης εάν δεν περιλαμβάνει και τις ποσοστώσεις. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου, ερχόμενες εβδομάδες έτσι και σε τεχνικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο αλλά κυρίως και πρωτίστως σε πολιτικό επίπεδο, το είπατε και εσείς, είναι κυρίως ε, μια ε, πολιτική πρόκληση. Ε, θα συνεχίσω λέω τις προσπάθειές μου έτσι ώστε να επιτύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που μου άρεσε στις παρεμβάσεις σας είναι επίσης τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία άκουσα σε σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες οι οποίες ε, ε, ήδη ε, εφαρμόζονται. Ναι, καλό θα ήταν να είχαμε μια οδηγία πλαίσιο πριν από 10 χρόνια η οποία θα είχε καθορίσει τα κατόφλια για τις διάφορες χώρες αλλά από την άλλη πλευρά ε, ήδη βλέπω ότι υπάρχουν πολλές χώρες και πολλοί σε το ε, διεπίστωσαν ότι υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει σχετικές με το θέμα νομοθεσίες Αλλά το σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει τα μηνύματα αυτά τα οποία θα ενθαρρύνουν τις χώρες που έχουν ξεκινήσει να προχωρήσουν και να οθήσει τις χώρες οι οποίες ακόμα είναι διστακτικές να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Πριν ολοκληρώσουμε ε, αυτήν την ε, συνεδρίαση ε, υπάρχουν δύο άτομα που θα κάνουν τις τελικές παρατηρήσεις, closing remarks. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Ζορντάν. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε για την δέσμευση την οποία δείξατε και την συνεκτικότητα των παρουσιάσεών σας που συνάδουν με την σημασία του θέματος. Ε, θα θέλαμε σήμερα πραγματικά δύο χρόνια μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου ε, σε πρώτη ανάγνωση, ε, δύο χρόνια μετά την κοινή θέση επί της οποίας συμφώνησαν οι πολιτικές ομάδες επί μιας αντικειμενικής θέσης που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Είναι δυτή η σημασία του θέματος. Έδειξαν ότι η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια καλύτερη διακυβέρνηση και καλύτερες οικονομικές επιδόσεις ε, και ε, η ερώτηση η οποία αντυχεί παντού είναι τι περιμένουμε έτσι ώστε να δώσουμε στις γυναίκες τις δυνατότητες να επιτύχουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους που μπορούν. Απ' την άλλη πλευρά ε, καταδεικνύει ότι η διοικητική πίεση μπορεί να λειτουργήσει, να δώσει αποτελέσματα. Μετά από δύο χρόνια έχουμε αύξηση περίπου της τάξης του 4% της παρουσίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, πράγμα που δείχνει ότι ε, νομοθετική πίεση μπορεί να έχει ε, θετικές επιπτώσεις, οι οποίες πλέον μετριούνται με τρόπο Επομένω, Επομένως, ε, τα νομοθετήματα αυτά, ε, το νομοθέτημα αυτό μπορεί να έχει ε, την αναμενόμενη επίπτωση στις ε, επιχειρήσεις οι οποίες θα θελήσουν να προλάβουν την ε, υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας. Εδώ έχουμε πλέον ένα κείμενο το οποίο μπορεί να ε, καθησυχάσει όσους προβληματίζονται. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι αυτός σκοπός αλλά είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη ενός σκοπού. Τώρα, εάν τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να αναλάβουν δεσμεύσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν και δεν έχουν τίποτα να φοβούνται γιατί όλα υπάρχουν μέσα στο κείμενο και περιλαμβάνεται και η περιβόητη ρήτρα ευελιξίας. Θέλουμε λοιπόν τώρα δέσμευση από τα κράτη-μέλη και συνοχή έτσι ώστε να επιτευχθούν αυτά αποτελέσματα. Φτάνω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μου σημείο για να υπενθυμίσω ε, ότι μπορούμε να έχουμε ένα εφέσιον βάδας ε, ε, ε, έτσι ώστε στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας όχι μόνο με τα παράλληλα μέτρα τα οποία μπορούν να έχουν καλά αποτελέσματα αλλά και σπάζοντας τους κώδικες που λειτουργούν, που ισχύουν αυτή τη στιγμή στα διοικητικά συμβούλια. Έφτασε η ώρα τα κράτη-μέλη να αγγίξουν το θέμα, να ασχοληθούν με το θέμα. Κυρία Υπουργέ, είμαστε στο πλευρό σας, σας στηρίζουμε. Ε, χαιρόμαστε που το θέμα αυτό εμφανίζεται πλέον και περιλαμβάνεται στη μέση διατάξη του Συμβουλίου τη 7 η Δεκεμβρίου. Ε, έχουμε, ε, ε, έχουμε εκατομμύρια Ευρωπαίων που περιμένουν ένα μήνυμα πιο συγκεκριμένο και θα πρέπει να δείξουμε όλοι το σθένος έτσι ώστε να προχωρήσουμε το θέμα μέχρι το τέλος γιατί είναι η, μόνη οδηγία η οποία πραγματικά αγγίζει την ισότητα ανθρώπων και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ και την πραγματικά τελευταία λέξη την πει η κυρία Γκρέγκρε. Ευχαριστώ. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όταν ψηφίσαμε για την έκθεση τη περασμένη θητείας... που είναι ήδη πριν από δύο χρόνια, έχει περάσει αρκετό καιρό, στην αρχή είχα φανταστεί, αμάν, θα βρούμε τον πελά μας με τις φεμινίστριε. Ε, και τώρα δούμε τι λέει η οδηγία. Ε, εντάξει, πρόκειται για τα διοικητικά συμβούλια εποπτικά συμβούλια με ευελιξία, όχι με αυστηρά κριτήρια και ποσοστώσεις. Και στις κυρώσεις τελικά πρόκειται για εργαλεία και μέσα που προτείνουμε και που ανταποκρίνονται και σέβονται απολύτως την αρχή της επικουρικότητας. Και δεν μπορούν να έχουν δικαιολογία τα κράτη-μέλη ότι τους επιβάλλει κάτι η Ευρώπη. Ε, δηλαδή ήταν μια ποσόστοση γυναικών light, ας πούμε, έτσι, μια ε, ελαφρά ρύθμιση για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την ισότητα στις εταιρείε. Και αντί να μας φυλάνε τα χέρια και να μας ευχαριστούν, ε, αρχίζουν και βάζουν διάφορα προσκόμματα και επιχειρήματα για τη δικαιοσύνη, για την ισότητα. Ε, συμφωνήσαμε με την οδηγία και κάναμε ένα δώρο στο Συμβούλιο, το οποίο τώρα κάθεται και το λιβανίζει αυτό το θέμα και αντέβεται. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μούτς για την ε, δέσμευσή σας και την επιστολή όμως που απευθύνατε μαζί με την Επίτροπο την κυρία Γιούροβα προς τους υπουργού γιατί καμιά φορά όταν ακούν οι υπουργοί ποσοστώσεις έτσι κάπως βγάζουν σπηριά. Τώρα όμως υπάρχει ένα καλό πνεύμα. Είναι light, επαναλαμβάνω, η πρόταση, πολύ ε, ε, ήπια και μπορεί να πείσει και τους πλέον συντηρητικούς. Τι άλλο να κάνουμε πια κι εμείς. Να στείλουμε επιστολές στους υπουργούς μας. Μπορεί να γίνει και αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν είναι κάθετα αντίθετοι, αλλά κάπως καλύπτουν τα νότα τους και ψιλοκρύβονται κτλ. Ε, να φροντίσουμε λοιπόν μέχρι το Δεκέμβριο και σε εθνικό επίπεδο να ε, παίξουμε μπάλα. Πολύ ωραία επιχειρήματα ακούσαμε από τον ΩΣΑ, πάρα πολύ χρήσιμα και διεξοδικά. Ξέρουμε δηλαδή ότι και οικονομικά δεν συμφέρει να μην έχεις γυναίκες. Και είναι και πώς να το πω, κάπως, με, κάπως, κάπως ε, μικρόψυχο, κάπως κακεντρεχές να μην ψηφίσει αυτή την οδηγία. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ενισχύεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια από την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν και φυσικά τους προσκεκλημένους ή τις προσκεκλημένες μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, δεν απομένει παρά να ε, καλέσουμε τους συναδέλφους των χωρών που δεν κατονομάστηκαν να κινητοποιηθούν και να σας ευχηθούμε κουράγιο, ε, πολύ ενέργεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία φυσικά κύριε Υπουργέ.